με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχουν ε, δώσει ενδείξεις για παραβίαση της συμφωνίας SWIFT. Γι' αυτό το λόγο δεν συμφωνώ με την αναστολή της συμφωνίας. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συναδελφοί, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία κυρία Ενφιάς. Ε, η, συζήτηση αυτή έχει ολοκληρωθεί. Να σας υπενθυμίσω ότι το σχετικό ψήφισμα θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλη, τη δεύτερη του Οκτωβρίου δηλαδή. Σημείο στην ημερήσια διάταξη, προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου ε, στην ΕΕ. Και θα δώσω πρώτα στο λόγο στο συντάκτη της προφορικής ερώτησης, τον συνάδελφο Λόπες Ακυγιάρ. Gracias, señora presidenta. De nuevo, todos Όλοι συμφωνούμε ότι το ιδιοσυνοριακό έγκλημα αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελική έκθεση της Επιτροπής ε, Κρίν το αναφέρει τα. Το ίδιο και η τελευταία αξιολόγηση ΣΟΚΤΑ της ε, αξιολόγησης των, ε, του σοβαρού και οργανωμένου κλίματος της Europol. το οργανωμένο έγκλημα λειτουργεί μέσω δικτύων σε διεθνές επίπεδο ε, σε πολλές χώρες ταυτόχρονα και σε πολλές περιοχές ταυτόχρονα. Ε, όχι μόνο παίρνουν εύκολα τα παλιά σύνορα, αλλά και υφίσταται και το γεγονός ότι ε, το έγκλημα δεν μπορεί να, να συνδεθεί με κάποιες συγκεκριμένες μόνο Αυτά τα εγκληματικά δίκτυα θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτελεσματική χρήση όλων των διασυνοριακών μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών και επιχειρησιακής συνεργασίας που διαθέτουμε. Η πρόκληση είναι τεράστια για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημερινή συζήτηση θα πρέπει να προσπαθήσει να συνεισφέρει στο πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε και να οργανώσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας για ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να εφαρμόζεται καλύτερα η, ευρωπαϊκή νομοθεσία και προκειμένου να ε, συλλαμβάνονται ε, οι εγκληματίες το συντομότερο δυνατό. Έχουμε ε, μια πανοπλία ε, εργαλείων για να συλλέξουμε, να επεξεργαστούμε και να συγκρίνουμε πληροφορίες και σε δικαστικό και σε αστυνομικό επίπεδο. Αλλά αυτά τα εργαλεία δεν ε, σχεδιάστηκαν εξ αρχή, Τα αναπτύσσουμε σταδιακά και μάλιστα πολλές φορές αλληλοεπικαλύπτονται ε, ή δεν τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά, ακόμα και ε, χωρίς διαφάνεια. Χρειάζεται λοιπόν ένα συνεπές και σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο όλα αυτά τα εργαλεία να αξιολογηθούν ταυτόχρονα και να χαράξουμε ένα χάρτη της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων. Μια αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση. Η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει ε, ένα όραμα για το μέλλον ε, που θα οδηγήσει σε μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις ε, προσπάθειες για να βελτιώσουμε και για να βελτιώσουμε την, ανταλλαγή, την καταπολέμηση του εγκλήματο, προστατεύοντας τα δεδομένα και τις ελευθερίες. Αναλογικότητα, διαφάνεια, ε, ε, κατά την ε, σύγκριση και την και, τον, και τη συλλογή πληροφοριών. Μην θυμηθείτε την απόφαση πριν το 2005, 7 κράτη-μέλη υπό την ομπρέλα της Επιτροπής ΠΡΙΜ είχαν ε, ξεκινήσει μια προσπάθεια αναζήτησης και αυτόματης ε, ε, σύγκρισης στοιχείων από βάσεις δεδομένων DNA, δακτυλικών αποτυπάτων κλπ. Ε, η απόφαση πριν ε, ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις αστυνομικές αρχές, αλλά θα πρέπει η πριν να λησβονοποιηθεί, λησαβονοποιηθεί. Γιατί τότε είχε, γίνει, είχε ληφθεί στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα που ήταν διακυβερνητικός. Οπότε δεν υφίστατο δημοκρατικός έλεγχος ε, ο οποίος πλέον έχει γενικευθεί μέσω της ενδείξης Λισαβόνας. Συνεπώς, ε, η Κομισιόν έχει σκοπό να προωθήσει την λισαβονοποίηση της απόφασης πριν. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σωστή ερμηνεία του πρωτοκόλλου 36 τη ε, ε, Συνθήκης Λισαβόνας. Θα ήθελα η Κομισιόν να λάβει αυτή τη δέσμευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη. Ε, πάνε ώρες που στέκομαι εδώ. Ε, ευχαριστώ και την Λίβε και τον πρόεδρό του που έθεσαν αυτό το θέμα. Όπως είπατε, η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την συνεργασία ε, την αστυνομική στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Καλωσορίζουμε τις αλλαγές της συνθήκης της Λισαβόνας και ε, κυρίως ε, αυτές που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στους τομείς αυτούς πλέον. Όσον αφορά την απόφαση ΠΡΟΥΜ, η Κομισιόν αποφάσισε να μην ε, ε, επιβάλλει αλλαγέ στην νομική βάση πριν έχουμε την πλήρη εφαρμογή. Διαφορετικά θα καθυστερήσει η εφαρμογή και θα καθυστερήσει όλη η διαδικασία σαν συνέπεια πιέζουμε για να γίνει η ταχύτατη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη σε ένα νομικά σταθερό περιβάλλον. Αυτό εγκρίθηκε αυτή η συμφωνία υπό τον τρίτο πυλώνα. Άρα η Κομισιόν δεν έχει τους ε, συνήθει ε, κανόνες για έλεγχο τη εφαρμογής ε, σε αυτή την περίοδο από το Δεκέμβριο όμω το 2014 μπορούμε να θέλουμε να κινήσουμε διαδικασία σε παραβάση. Έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζονται νέα ευρωπαϊκά εργαλεία ανταλλαγή πληροφοριών αυτή τη στιγμή. Τα υπάρχοντα εργαλεία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο και κάνουμε συγκεκριμένε συστάσει γι' αυτό. Παραδείγματο χάρη να συμφωνήσουμε για ένα κοινό κανάλι επικοινωνία, ε, κατά προτίμηση μέσω τη Europol, να υπάρχει ένα ε, σημείο επαφή ε, ανακράτω για να ανταλλάσσονται αυτέ τι πληροφορίε για τα διασυνορικά θέματα και να γίνεται συνεχώ κατάρτιση για την χρήση αυτών των εργαλείων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υψηλά επίπεδα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων και στατιστικές αξιόπιστες. Ε, η συζήτηση για το πώς θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εργαλείων, καναλιών κλπ. Ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι κάτι που συνεχίζεται εδώ και αρκετό καιρό και ε, έχουμε εμπνευστεί και από την δημοσίευση της ε, ανακοίνωσης και η συζήτηση αυτή γίνεται τώρα σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλέ φορέ με του υπουργού έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά και πιέζουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με την εφαρμογή. Τέλο, για την προστασία των δεδομένων, θα ξέρετε βέβαια ότι η προτινόμενη οδηγία για την ε, προστασία των δεδομένων περιλαμβάνει δέσμευση εκ μέρου τη Κομισιόν να επανεξετάζει τα υπάρχοντα νομικά μέσα ε, στον τομέα αυτό ε, τρία χρόνια από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία. Αυτά προ το παρόν, αλλά βεβαίω περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε και τι προτάσει σα. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτον, ο κύριος Δίας Δεμέρα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, επίκαιρη η προφορική αυτή ερώτηση, η οποία μου βρίσκει σύμφωνο. Ε, η καταπολέμηση του διασυνορικού εγκλήματος είναι περίπλοκη και αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στην εντατικοποίηση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για ποινικά δικήματα. Το 2005 ε, υπογράφηκε η συμφωνία Πρίμαν μεταξύ 7 κρατών μελών ε, που τελικά ευθύθηκε το 2008. Η επιτυχία της ε, οδήγησε σε πολλά άλλα κρατημέλη να θέλουν να συνδεθούν. Κάτι που την έκανε κοινοτικό εργαλείο όμως ε, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρόμοιες αρμοδιότητες σε αυτά τα θέματα, ε, οι διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες των κρατών μελών, καθώς επίσης και η ύπαρξη διαφόρων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, ΣΥΣ, συς 2 κλπ. Ε, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πανόραμα πολύ περίπλοκο που δεν διευκολύνει την συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά Συμφωνώ με τα συμπεράσματα της ε, Κομισιόν στην ανακοίνωση της 7ης Δεκεμβρίου. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες βάσεις νέα εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών. Αντιθέτως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία ε, πιο αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο η νομοθεσία να προσαρμοστεί συνθήκη της ε, Λισαβόνας με περισσότερες εγγυήσεις και να τεθεί σε δημοκρατικό έλεγχο. Η Λισαβόνα θα πρέπει να αντικαταστήσει μια απόφαση του τρίτου πυλώνα, χωρίς να ξεχνάμε τις βασικές αρχές της αρχικής συνθήκης πριν. Προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου και ιδιαίτερα στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των ατομικών δεδομένων ε, και οποιοδήποτε περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων ε, θα ε, πρέπει να γίνεται δεκτός μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η απόφαση πριν είναι και αυτό. Συγχαρητήρια. Gracias, señor Díaz frau präsidentin! Συμφωνώ με την εκτίμηση του κ. Διαστεμέρα για την ε, Συμφωνία Προυμ. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και μαζί με ε, και δίνει στι αρχέ στι δικαστικέ και τι αστυνομικέ ένα πολύ σημαντικό μέσο κατά πολέμη εγκληματικότητα. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να προφυλάσσονται και να διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα. Στη συμφωνία αυτή δυστυχώ όμω υπάρχουν πολύ σημαντικέ αδυναμίε ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα γιατί δεν υπάρχει καν ορισμό των προσωπικών δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια από το 2008 έχει τοποθετηθεί με μια γνωμοδότηση και έχει ζητήσει τον ορισμό των προσωπικών δεδομένων, αλλά και η σύμβαση του 1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μιλάει για προσωπικά δεδομένα δίνει επαρκή ορισμό και ορίζει αυτά τα προσωπικά δεδομένα ως υποκειμενικά δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και την απαγόρευση της διάθεσή του σε μη ε, αρμόδιες αρχές. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι ο κανονισμός, ε, η σύμβαση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, είναι πολύ σημαντική όπως και η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα, αρκούσαν, να αξιοποιούνταν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. θα ήλπιζα δε πώς είχαν δείξει πολύ, μεγάλη, ε, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στην ε, εφαρμογή της ε, σύμβασης Πριμ, μάλλον στην υπογραφή της πριν από τέσσερις εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνα της συνθήκης σύμβασης Πριμ, να είχαν δείξει οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις αντίστοιχο ενθουσιασμό και για τον ορισμό των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με χαρά σας βλέπω εδώ. Ξέρω ότι έχετε μόλις γύρισε από τη Λαμπεντούσα, ξέρω ότι ζήσατε ε, στον απόϊχο μιας μεγάλης ε, τραγωδίας. Εδώ τώρα καλούμεθα να μιλήσουμε για ασφάλεια και ξέρουμε ότι τα σύνορά μας δεν αποτελούν πλέον ε, επαρκή προστασία για τον πολίτη της Ευρώπης. Αυτό γνωρίζει και ο ίδιος ο πολίτης. Μετά μιλούμε για την ανασφάλεια ως προς την οικονομία, ως προς την οικονομία και την απασχόληση. Μιλάμε όμως επίσης και για την υπερσυνοριακή οργανωμένη εγκληματικότητα που έχει πολύ μεγάλη σημασία και που αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για συνεργασία. Ένας κοινό λοιπόν ορισμός της οργανωμένης διασυνοριακή εγκληματικότητα ε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. είτε πρόκειται για πορνεία είτε πρόκειται για ε, λαθρεμπόριο όπλων είτε για λαθρεμπόριο ναρκωτικών έχουμε να κάνουμε με τεράστια προβλήματα με εκατομμύρια σε οικονομικού όρου και βλέπουμε ότι οι διακινητέ, σε παραδείγμα στη Λαμπεντούζα δεν οροδιούν προ και θέτουν σε κίνδυνο τόσε ανθρώπινε ζωέ. Πρέπει τώρα λοιπόν να πιέσουμε ώστε να λειτουργεί η υγιής ή νόμιμη οικονομία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καλά μέσα, επικοινωνία, πληροφορίες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Στη δική μου την ιδιαίτερη πατρίδα μάλιστα πρέπει να πω ότι αναπτύσσονται κάποιες ανταλλαγές πληροφοριών πέραν των συνόρων οι οποίες έχουν αποδώσει άριστα αποτελέσματα. Και γι' αυτό δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι τόσα τα κράτη-μέλη που διστάζουν να προχωρήσουν σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών γιατί τελικά ο μόνος ο οποίος κερδίζει από την ε, άρνηση κρατών μελών να διαθέσουν στοιχεία τους είναι ο εγκληματίας, η εγκληματική οργάνωση. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει αποφασιστικά. Χρειάζεται ένα ευρύ ευρωπαϊκό πλαίσιο, ε, ενισχυμένη Europol, ενισχυμένη και ισχυρή Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται τον άλλο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φράξει το δρόμο στον οργανωμένο εγκληματία. Χρειάζεται λοιπόν βεβαίως να γίνεται σεβαστή η, ε, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το απόρριτό του, αλλά πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει και την ασφάλεια για τους πολίτες μας. Ο κύριος Άλμπρεχτ εκ μέρους των Πρασίνων. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εκφραστώ ως εξή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλύτερη συνεργασία για την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές στην Ευρώπη Ευρώπη, είναι απαραίτητο, αλλά το δήλωσε και το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια, το δηλώνει η ομάδα μου. Χρειαζόμαστε κοινέ προδιαγραφέ για την καλύτερη αυτή συνεργασία. Κοινέ προδιαγραφέ όταν έχουμε να κάνουμε την προστασία των δεδομένων, όταν έχουμε να κάνουμε με τα δικονομικά δικαιώματα, όταν έχουμε να κάνουμε τι αρχέ του δικαίου, του κράτου δικαίου, αρχέ που είναι εγγεγραμμένε στα συντάγματά μα. Δεν αρκεί να λέμε αμοιβαία αναγνώριση των κοινών προδιαγραφών στην Ευρώπη. Δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Α δουλέψουμε πάνω στι κοινέ προδιαγραφέ και μετά να διευκολύνουμε το έργο των δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Και επίση, δεν θέλω να συμπληρώσω, πρέπει να εστιαστούμε στα μέσα εκείνα τα οποία πράγματι διευκολύνουν τη συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην περιοχή που αυτό χρειάζεται και όχι να διαθέτουμε εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για συστήματα παρακολούθησης και επιτήρησης τα οποία εν τέλει δεν έχουν αποδειχθεί κατά την άποψή μου και τόσο αποτελεσματικά δεδομένου ότι πολύ λίγα εγκλήματα εξηχνιάζουν αλλά βέβαια καλό θα είναι να ενισχύσουμε τις δυνάμεις σε προσωπικό της Europol και τον συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο, σε μικρή κλίμακα. Εκεί ακριβώ χρειάζεται να κάνουμε δουλειά, αλλά δυστυχώ δεν είναι αυτή η πρόθεση και η διάθεση των κρατών μελών και του Συμβουλίου και από ό,τι φαίνεται ούτε εσεί, ούτε εσεί, κυρία Επίτροπε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση. Κύριε Οι εθνικές ε, αρχές ε, πρέπει να συνεργαστούν, να συνεργάζονται για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα κανάλια συνεργασίας. Γι' αυτό λόγο χρειαζόμαστε κοινέ προδιαγραφές σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως εισηγήτρια για τον κανονισμό Eurodac ε, γνωρίζω πόσο οι, πώς λειτουργούν οι ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων Eurodac επιτρέπει ε, την πρόσβαση στις εθνικές αρχές προκειμένου να προλάβουν τρομοκρατία και σοβαρά εγκλήματα και για να προστατέψουν μάρτυρες. Ε, οι ερευνητές μπορούν μέσω αυτών των στοιχείων ε, να ελέγξουν το κατά πόσον ε, το οργανωμένο έγκλημα προσπαθεί να εισάγει μέσα στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέλη του με ψευδή στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σύστημα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Όμως τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, για, ε, στην Eurodac αν δεν ε, ψάξουν τα ίδια στοιχεία στην βάση δεδομένων πριν, που όμως υπάρχει μόνο σε 11 κράτη-μέλη. Συνεπώς περιορίζεται η πρόσβαση. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει όλα την συμφωνία πριν και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Θα πρέπει η Κομισιόν να τα πιέσει προκειμένου πράγματι να βελτιωθεί η καταπολέμηση του διασυνορικού εγκλήματο. Δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Βάντενκαμπ. Κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει ένας τομέας στην Ευρώπη που πραγματικά καταλαβαίνει τη σημασία των ανοιχτών συνόρων και τη ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι το οργανωμένο έγκλημα. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μου, στις κάτω χώρες, με τα ανοιχτά σύνορα. Νομίζω ότι σε ορισμένα ζητήματα ε, πραγματικά ε, δεν κατανοούμε ε, τι παίζεται. Πολύ πρόσφατα συνελήφθη ένας νέος μαφιόζος που για πολλά χρόνια ε, ζούσε σε ε, ένα διαμέρισμα δημόσια χωρίς να τον αγγίζει κανείς μέχρι ε, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων. Έτσι τον εντοπίσαμε. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η ανταλλαγή στοιχείων στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Η ερώτηση είναι εξής. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η εφαρμογή πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι μόνο 11 κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει την συμφωνία πριν. Γιατί οι υπόλοιπε χώρε δεν ακολουθούν. Συμφωνώ με τον κύριο Αγγιλάρ επίση ότι χρειάζεται και δημοκρατικό έλεγχο ε, της καταπολέμησης αυτού του εγκληματο. Η Κομισιόν ε, είπε ότι θα προβεί σε δημοκρατικό έλεγχο όταν όλοι έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Πότε θα γίνει αυτό, πόσο θα περιμένουμε ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά από τα προβλήματα που έχουμε στην Ένωση είναι η μη ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένα πραγματικό δημοκρατικό έλλειμμα και ελλειπή έλεγχο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μια χαρτογράφηση λοιπόν των εθνικών νομοθεσιών, των διεθνών συμφωνιών που εμποδίζουν το, τη διασυλλογική ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει επίση η Κομισιόν να αυτοματοποιήσει τι διαδικασίε για την εφαρμογή των υπαρχόντων συστημάτων για να υπάρχει ένα ενιαίο φόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσταθούν και μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ε, εκπαίδευση της αστυνομίας για να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία. Τέλος, ε, ένα εργαλείο που ε, συνηθίζεται στην ανταλλαγή, στη συνεργασία των αστυνομιών. Πρέπει απλώς να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δώσουμε καλύτερες απαντήσεις στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ κύριε Σκούρια. Προχωρούμε με τη διαδικασία Catch the Eye και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λούχαν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε πάντα για προστασία δεδομένων. Διαφάνεια και πολλά βέβαια λέγονται και από την άλλη πλευρά ότι θέλουμε και πιο πολλέ πληροφορίε και ενημέρωση, ανταλλαγή στοιχείων για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το έγκλημα αλλά και να εξασφαλίσουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία. Αλλά κοινέ προδιαγραφές δεν μπορούμε να αναπτύξουμε. Δεν είμαστε σε θέση να συντονίσουμε τις ε, δεν μπορούμε να συντονίσουμε τις αρχές μας. 17 κράτη εκπροσωπούνται με εμπειρογνώμονες, με στοιχεία που θα πρέπει να διατίθενται κατά τρόπο διαφανή και με σεβασμό της ασφάλειας των πολιτών. Η κατάσταση είναι καταστροφική βέβαια σε, πολλά, σε πολλούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και στη σχέση μεταξύ των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε καλύτερη εστίαση. Για όποιο σύστημα και να μιλάμε, για το ΣΥΣ, για το Eurodac, για οτιδήποτε πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. Ευχαριστώ. ja osobiście jestem zdania bardzo dobrze, że o to pytamy, bardzo dobrze, że o to rozmawiamy. Dlaczego? Jednym z... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ θετικό το ότι κατατέθηκε αυτή η προσωπική ερώτηση, η προφορική ερώτηση, συγγνώμη, γιατί πρέπει να δείξουμε ότι τηρείται όπως πρέπει στους όρους που πρέπει το νομοθέτημα αυτό και όταν παραβιάζεται δεν επιτρέπεται καμία ατιμορρησία. Δεν επιτρέπεται καμία ατιμορρησία και ε, πρέπει κάθε διασυνοριακή εγκληματική δραστηριότητα να ανοιχνεύεται ώστε να καταπολεμείται αποτελεσματικά το έγκλημα. Το μόνο μέσο που έχουμε λοιπόν στη θέσή μας είναι το πιο σημαντικό, είναι αυτό το μέσο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για να κερδίσουμε και το σεβασμό των πολιτών μας. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τα, τους ευρωβουλευτές για τα, τις απόψεις τους. Ε, είναι πραγματική πρόκληση το διασυνορικό έγκλημα. Ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι η πιο στενή συνεργασία των ε, υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Γι' αυτό τον ε, λόγο ε, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή καινούργια εργαλεία, καινούργιες ιδέες ανταλλαγής πληροφοριών. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε ήδη. Μόνο τα μισά μέλη έχουν πράγματι εφαρμόσει την απόφαση πριν. Οπότε δεν έχει νόημα να αλλάξουμε την νομική βάση. Γιατί καθυστέρηση. Προσπαθούμε να, να το απαντήσουμε κι εμεί. Σε ορισμένε περιπτώσει είναι πρακτικό το πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη δεν ξέρουν πώ. Γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτούμε μαθήματα και εκπαίδευση. Επίση, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν το ένα το άλλο. Αυτή είναι κυρίω η λόγη τη καθυστέρηση. Τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν και βέβαια δεν είναι και πρώτη προτεραιότητα. Όμω προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε και πολλέ συναντήσει του Συμβουλίου Τζάι. Έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ε, εντείνουν τις προσπάθειές τους. Πότε θα καταλήξουν αυτές τι προσπάθειες. Δεν μπορώ να σας πω ότι σε ένα χρόνο θα έχει λησαβονοποιηθεί πλήρως. Ελπίζω σε ένα χρόνο να την έχουν, έχουν εφαρμόσει, να έχουν εφαρμόσει την απόφαση πριν όλα τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε κοινέ προδιαγραφέ, χρειαζόμαστε να δούμε και την προστασία των δεδομένων. Και μόλι η εφαρμογή προχωρήσει, θα ξεκινήσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για περαιτέρω βελτίωση συνεργασία. Στο πλαίσιο της ε, Στοκχόλμης πάντοτε. Ε, λίγη συζήτηση, ευχαριστούμε Επίτροπε. Η ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το